special meeting. Καλησπέρα σας. Είναι μια τακτική συνεδρίαση, αλλά είναι η τελευταία μας φορά, η τελευταία φορά που θα συναντηθούμε επισήμως κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής ε, θητείας. Πολλοί συνάδελφοι που έχουν ήδη μπει σε ρυθμούς προεκλογικής εκστρατείας θεώρησαν ότι δεν θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Υπάρχουν όμως κάποιοι συνάδελφοι που είναι παρόντες. Οπότε να σας καλωσορίσω, να σας καλωσορίσω και όλους όσους μας βλέπουν από το διαδίκτυο. Είναι περίεργη αίθουσα. Σας βλέπω εκεί στο, βάσο, στο βάθος. Ξέρω ότι είναι και μια ομάδα επισκεπτών ε, του της περιφέρειας του Τόμας Μάν, αν δεν κάνω λάθος. Α, ναι. Το ξέρω πολύ καλά τον Τόμας Μάν. Είναι πολύ καλός ε, συνάδελφος, επιτροπής ε, απασχόλησης όμως, όχι της δικής μας επιτροπής. Ε, καλώς ήρθατε λοιπόν στην σημερινή μας συνεδρίαση. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει όλα, όλη την ομοθετική και μη νομοθετική μας δουλειά για την κοινοβουλευτική αυτή θητεία. Δεν έχουμε άλλες συζητήσεις λοιπόν σήμερα το απόγευμα. Επειδή όμως είχαμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, καλέσαμε επιτρόπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε πολύ στενά για την ολοκλήρωση σημαντικών νομοθετικών κειμένων. Τους καλέσαμε λοιπόν να έρθουν να μας ε, παρουσιάσουν τη δουλειά τους και τις εμπειρίες τους, ε, ίσως και κάποια διδάγματα ε, εν ώψη της μελλοντική μας δουλειάς, ίσως και κάποια εκρεμή θέματα που δεν ολοκληρώσαμε ακόμη. Υπάρχει ένα σημαντικό νέο ε, θέμα ε, το οποίο δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε, δεν μπορέσαμε να το συζητήσουμε καν σε αυτήν την κοινοβουλευτική θετία. Θα το κάνουμε λοιπόν στην επόμενη. Τέσσερις η ώρα θα ψηφίσουμε. Χαίρομαι που ο εισηγητής Κορέντε Κάμπος είναι εδώ είναι ο εισηγητής μας ε, για τον ε, προϋπολογισμό. Πρέπει να εγκρίνουμε μία επιστολή για την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ο κύριος ε, Μίμητσα, ο οποίος ήθελε να είναι εδώ σήμερα, γιατί ήθελε να μας παρουσιάσει και μία έκθεση την οποία ενδεχομένως να έχετε για την πολιτική για τους καταναλωτές. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα. Οπότε, στις 4 παρα 10 θα κάνουμε ένα διάλειμμα για τσάι, γιατί στις 5 θα έρθει ο Μισελ Μπαρνιέ να μας ε, παρουσιάσει εκείνος τον απολογισμό της δουλειάς του. Οπότε μετά τις 5 παρα 10 που θα κάνουμε το ε, διάλειμμα, Ελπίζω να είστε πίσω γέρος για να ακούσουμε τον ε, κύριο Μπαρνιέ. Είναι εδώ και συνάδελφοι, άλλοι εκπρόσωποι από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε το τέλος των εργασιών μας και την πολύ επικοδοματική συνεργασία μας. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει και το τελευταίο newsletter μας, το τελευταίο ενημερωτικό μας ε, δελτίο. Έχει και ένα μικρό ε, μήνυμα ε, από δικής μου πλευράς στο εξώφυλλο να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την, την ομάδα σύνταξης και όλους τους συνεργάτες του ενημερωτικού δελτίου. Βλέπετε ότι υπάρχει και ένα λευκό κομμάτι ε, στο κάτω μέρος της, ε, ε, του ενημερωτικού δελτίου για να μπορέσετε να συλλέξετε υπογραφές για σουβενίρ. Εγώ ήδη έχω βάλει τον κύριο Σεμέτα και έχει υπογράψει στο δικό μου. Αυτά ήθελα να σας πω. Να εγκρίνουμε επισήμως την ημερήσια διάταξη πριν δώσω το λόγο σε κάποιον άλλον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτε άλλο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, πρακτικά προσέγγιση; Α, υπάρχουν τελικά. Τα έχετε στο φάκελό σας. Πρέπει μέχρι το τέλος συνεδρίασης ε, ή μετά το κοκτέιλ, αν μπορείτε ακόμη, μετά το ποτό, να μας πείτε ότι συμφωνείτε με τα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής. Κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. μην είναι η τελευταία συνεδρίαση της οποίας προεδρεύεις γιατί θα συνταξιοδοτηθείς. Ε, παρά το γεγονός ότι ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες, θα ήθελα να πω ε, ότι εκτιμούμε όλους ιδιαίτερο το έργο σου. Ήσουν εξαιρετικός ε, ε, πρόεδρος, ε, άκουγε τις απόψεις όλων ε, και νομίζω ότι είναι πραγματικά υπόδειγμα η Επιτροπή μας. Νομίζω ότι και άλλες Επιτροπές θα έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Είναι η τελευταία σου συνεδρίαση, είναι η τελευταία σου ημέρα ως Προέδρου. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δουλειά σου. Λυπάμαι που δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι συνάδελφοι να εκφράσουν και εκείνοι τις ευχαριστίες τους, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική σου Προεδρία. Ο κύριος Μάντερς. Και εγώ να σου πω ε, μπορώ λοιπόν να σε καλέσω στην ε, ε, οικονομία των γκρίζων μαλλιών, για να το πούμε έτσι. Right. Good. No other, uh, will be, I'm sure, chance for... Um... Κύριε Σφάμπ, δεν έχετε τίποτα να μας πείτε για την ώρα. Ε, ίσως να έχουμε και την ευκαιρία στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μετά λοιπόν από την εισαγωγή αυτή που ήταν ιδιαίτερη γιατί είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα και λίγο περίεργη, να δώσω το λόγο στον Επίτροπο και να καλωσορίσω και μέλη της ομάδας του με τους οποίους ε, έχουμε συνεργαστεί πολύ και ειδικότερα τον κύριο Ζαλίσκι, γιατί τον έχουμε δει πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους στην Επιτροπή μας, ε, γιατί ήταν επικεφαλής της ομάδας σας για τον τελωνιακό κώδικα, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, τουλάχιστον από πλευρά τροπολογιών και εκτελεστικών πράξεων. Ελπίζω να συνεχιστεί η ηγεσία σας για το θέμα αυτό. Υπήρξαν και άλλα προγράμματα για τα οποία δουλέψαμε με εσά, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ε, στα τελωνία και γενικότερα τα θέματα που αφορούν ε, στα τελωνία. Με την υποστήριξή σας ε, και τη δική σας ε, ενημέρωση καταφέραμε να επισκεφθούμε πολλά τελωνία σε όλο τον κόσμο, στην Ινδία και στην Κίνα μεταξύ πολλών άλλων, όπως επίσης ε, και στην Κωνσταντινούπολη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε με τις επισκέψεις μας αυτές όλα αυτά ε, τα οποία κάνατε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ανοίξουμε και τον κατάλογο των ομιλητών για όλους όσους θέλουν ε, να σας ε, θέσουν ερωτήματα. Όχι, απλώ εκφράζει συμμετοχή στον κατάλογο ομιλητών. Σε ευχαριστώ, Μάλκομ, για τα σοβιακά σου αυτά λόγια. Καλησπέρα σε όλους, αξιότιμα μέλη και σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συνεδρίαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίδεται σήμερα η ευκαιρία να κάνω έναν απολογισμό των όσων έχουμε επιτύχει μαζί στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Μάλκομ ότι όντως έχουμε πετύχει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας και θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα αυτά. Στην αρχή της θητείας, το 2010, ο κόσμος βρισκόταν σε πολύ δεινή κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το νέο Κολέγιο των Επιτρόπων αντιμετώπιζαν πολλές προκλήσεις το θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινό θεματολόγιο για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνονταν περισσότερο στην ανάγκη να ανακάμψουμε από την κρίση και να καταφέρουμε να πετύχουμε μια κάποια οικονομική ανάπτυξη. Δεν έχουμε βγει ακόμα από τη δινή αυτή κατάσταση, αλλά μπορώ πραγματικά να πω ότι έχουμε πετύχει πολύ σημαντική πρόοδο από τότε. Μιλώντας τώρα εξ ονόματος ε, της ε, δικής μου της ε, θέσης, χαίρομαι πάρα πολύ για τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε πετύχει και τα επιτεύγματα αυτά δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα σήμερα θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την πολύ επικοδομητική και καρποφόρα συνεργασία που είχαμε με την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Θα ήθελα να κάνω μία σύντομη ανασκόπηση των σημαντικότερων επιτευγμάτων για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο. Τελωνία, καταπολέμηση της απάτης και φορολογία. Καταρχάς, κάποια σχόλια στον αφορά τον τομέα των τελωνίων. Οι αποτελεσματικέ και ομαλέ εμπορικέ ροέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα όμω θα πρέπει να έχουμε και ένα αποτελεσματικό έλεγχο για τι αλυσίδε εφοδιασμού και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε του σχετικού κινδύνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την ασφάλεια τόσο για την Ευρώπη όσο και για του καταναλωτέ τη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα τη εσωτερική αγορά Ευρωπαϊκή Ένωση από το παράνομο εμπόριο και το λαθρεμπόριο και την απάτη. Ως προς αυτά λοιπόν έχουμε κάνει έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο. Έχουμε βελτιώσει τους ελέγχους καθώς επίσης και τις εμπορικές ροές και αυτό χάρη στη δική σας την Επιτροπή. Ο Ενωσιακό Τελωνιακό Κώδικα αποτελεί μια πολύ σταθερή βάση προκειμένου να έχουμε ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό ηλεκτρονικό περιβάλλον για τα τελωνία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερω τη Σιλβάνα Ράπτη, τον Όλε Σμιτ και την Χάιντε Ρούλε. Και όλου ιδιαίτερω να ευχαριστήσω και την Κωνστάνσε Λεγκρίπ και βέβαια και εσά, Μάλκομ. Όλοι σας εργαστήκατε πολύ επικοδομητικά με το Συμβούλιο και από κοινού καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο για να συνδυάσουμε από τη μια την ασφάλεια και από την άλλη τη διευκόλυνση του εμπορίου για τους αξιόπιστους εμπόρους. Όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση για την κατάσταση της Τελωνιακή Ένωσης του 2012, η ολοκλήρωση του εξυγχρονισμού της Τελωνιακή νομοθεσίας αποτελούσε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια ισχυρή και ενοποιημένη τελωνιακή ένωση μέχρι το 2020. Η έγκριση λοιπόν του τελωνιακού κώδικα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ρώσιμο και μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Βέβαια πρέπει ακόμα να καταβληθούν προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή του κώδικα αυτού. Αλλά πλέον τώρα με την συνεργασία των κρατών μελών έχουμε θέσει και τα νέα βήματα τα οποία πρέπει να πετύχουμε στο μέλλον. Η ε, σταδιακή βαθμιαία προσέγγιση που προτείνει ο κύριος Ματέος Σαλβίνη στην έκθεσή του θα συνεχιστεί. Και να ευχαριστήσω επίση και τον Ραφαέλε Μπαλτασάρε για τι δικέ του τι προσπάθειε όσον αφορά την έγκριση του προγράμματο Τελωνία 2020. Το βασικότερο αυτό κοινοτικό μέσο για την υποστήριξη του εξεχρονισμού έχει πλέον υιοθετηθεί. Μια άλλη προτεραιότητα την οποία θέσαμε στην ανακοίνωση του 2012 ήταν η αναθεώρηση της υφιστάμενης διακυβέρνησης της Ελληνικής Ένωσης και αυτή η διεργασία έχει ξεκινήσει. Το τρέχον αποκεντρωμένο σύστημα για την εφαρμογή και τη διαχείριση της Ελληνικής Ένωσης παρουσιάζει βέβαια κάποιες αδυναμίες, για παράδειγμα όσον αφορά την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας και όσον αφορά τις περιτές και δαπανηρές επικαλύψεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Το Μάρτιο του 2014, οι γενικοί διευθυντέ των 28 Τελωνιακών αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν μεγαλύτερη αντιστοίχηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την εφαρμογή τη ελληνική νομοθεσία. Είπαν επίση ότι θα πρέπει να αυξηθεί το πολιτικό προφίλ των τελωνίων, καθώ επίση και των υπηρεσιών που παρέχουν τα τελωνία προ την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους ερχόμενους, λοιπόν, τους ερχόμενους μήνες θα παρουσιάσουμε ένα νέο προσχέδιο για την περίοδο μετά από το 2020. Θα παρουσιαστεί το προσχέδιο αυτό στα τέλη της δικής μου θητείας. Η επόμενη όμως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θέσουν υψηλά τον πύχη της φιλοδοξίας. Και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε ανάλογα αποτελέσματα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα τελωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή όσον αφορά το παγκόσμιο προσκήνιο. Όσον αφορά τώρα τους διεθνεί μα εταίρου, σημαντικέ προσπάθειες έχουν καταβληθεί για να προωθήσουμε εταιρικέ σχέσει και συνεργασίε με τι όμορε μα χώρε, καθώ επίση και με του διεθνού μα εταίρους. Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε ιδιαίτερα την τελωνιακή συνεργασία με τι τρίτες χώρε και έχουμε καταφέρει κατά αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε και να συμπληρώσουμε τι προσπάθειε που γίνονται στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καταφέρει να διευκολύνουμε περισσότερο το εμπόριο, καθώς επίσης και να επιβάλλουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με τους βασικούς μας εταίρους, δηλαδή τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία. Επίση, η προσέγγιση συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπω φαίνεται ιδιαίτερα μέσω τη έννοια του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, αρχίζει και επεκτείνεται όλο και περισσότερο προ του εμπορικού μα εταίρου. η αξιόπιστοι εμπόρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρουν πλέον ενό καθεστώτο αμοιβέ αναγνώριση με βασικού μα εταίρου όπω η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ελβετία και η Νορβηγία. Ελπίζω θα καταφέρουμε να έχουμε καθεστώ αμοιβέ αναγνώριση πολύ σύντομα και με την Κίνα. Όσον αφορά τι πολυμερεί μα σχέσει, η ολοκλήρωση τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη διευκόλυνση του εμπορίου στο Μπάλι αποτελεί μια πολύ σημαντική νίκη για μα. Καταδεικνύει πλέον ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για τα τελωνία παγκοσμίω τα ευρωπαϊκά τελωνία μπορούν και θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, θα έχουν ηγετική θέση. Παράλληλα με τη διευκόλυνση του εμπορίου, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ πλέον να πω ότι παρέχουμε καλύτερη προστασία και προστατεύουμε τόσο τους πολίτες όσο και την εσωτερική αγορά, καθώς επίσης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προφανώ τα τελωνία διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να μην φτάνουν στην εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση παραποιημένα προϊόντα, προϊόντα απομίμηση. Η επιβολή λοιπόν των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη, αλλά και όλου ιδιαίτερου για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο. Και βλέπω ότι το ζήτημα αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργεν Κρότσμαν, για τις προσπάθειες οι οποίες κατέβαλε προκειμένου να εγκριθεί ο κανονισμός για την επιβολή, την τελειωνιακή επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Μέσω του νέου αυτού κανονισμού έχουμε καταφέρει να αποσαφηνίσουμε τις διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούμε και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε ακόμα και τα μικρά φορτία προϊόντων στον πιο προβληματικό τομέα, ο οποίο είναι οι πωλήσει μέσω του διαδικτύου. Έχουμε καταφέρει να έχουμε καλύτερη προστασία τόσο για του πελάτε, του καταναλωτέ, όσο και για του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Επίση, έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα τη πρόσβαση στα φάρμακα. Το ζήτημα αυτό έχει πλέον επιληθεί. Χαίρομαι επίση που σα λέω ότι ο σχετικό κανονισμό όχι μόνο υποβλήθηκε, προτάθηκε, αλλά καταφέραμε να τον διαπραγματευτούμε και να τον εγκρίνουμε κατά τη διάρκεια τη δική μα θητεία και ήδη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Και έχουμε επίση και τη βάση δεδομένων κόπη, η οποία διασυνδέει όλα τα κράτη-μέλη και αυτή λειτουργεί πλήρω. Με την έγκριση του νέου κανονισμού για την τελειωνιακή επιβολή των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να θέτει, συνέχισε μάλλον να θέτει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά το διεθνές επίπεδο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και βλέπουμε ότι τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Κινέζοι φίλοι μας προσπαθούν να εμπνευστούν από τον δικό μας τον κοινοτικό κανονισμό. Σε προηγούμενε παρουσιάσει που έκανα στην Επιτροπή σα, αναφέρθηκα και σε πρωτοβουλίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των προϊόντων. Το ζήτημα αυτό μα απασχόλησε ιδιαίτερα σε συνεργασία με άλλε αρχέ αλλά και με τον εμπορικό κλάδο. Εφαρμόζουμε τώρα πλέον το πολιετέ σχέδιο δράση για την εποπτεία των προϊόντων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των συνοριακών μας ελέγχων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές θα καταφέρουμε να χαρτογραφήσουμε τι διαφορέ που υπάρχουν από τη μία χώρα στην άλλη όσον αφορά του συνοριακού ελέγχου και πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε πλήρω όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται στου ελέγχου αυτού. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα και όλου ιδιαίτερω την Κριστέν Σάλτελμον και τον Γιούργεν Κρόιτσμαν, οι οποίοι υποστήριξαν την ομάδα εμπειρογνωμόνων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εργάστηκε για τα ζητήματα επιτήρηση και βελτίωση των ελέγχων στα σύνορα. Εν τελευταία τέσσερα χρόνια καταφέραμε να εφαρμόσουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία την συστηματική ηλεκτρονική διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά τα τελωνία. Καταφέραμε επίσης να εγκρίνουμε την λεγόμενη Security Amendment, την τροπολογία για την ασφάλεια, η οποία απέτησε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά καταφέραμε τελικά να την εγκρίνουμε. Και θεωρώ πλέον ότι μπορούμε να αντλήσουμε από όλη αυτή την εμπειρία κάποια πολύ θετικά διδάγματα. Ο παγκόσμιο εντομισμό των κινδύνων και των επικίνδυνων προϊόντων, τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξακολουθήσει να, να αποτελεί προτεραιότητα και τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι μειώνονται όλο και περισσότερο οι σχετικοί εθνικοί προπολογισμοί, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε αποτελεσματική χρήση των κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Σύμφωνα με τι προτεραιότητες που έχουμε στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση των, της Ένωση, Ένωσης, έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε του κινδύνου ε, κινδύνους οποίου πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τον ε, Ιανουάριο του 2013 καταφέραμε μέσω της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαχείριση των κινδύνων να αντιμετωπίσουμε όλα τα κενά τα οποία υπάρχουν στην κοινοτική νομοθεσία και όλες τις αδυναμίες. Πολύ σύντομα, του επόμενου μήνε θα έχουμε ένα νέο σχέδιο δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος προτάθηκε μία οδηγία όσον αφορά την καταπολέμηση των τελεινιακών παραβιάσεων και τις σχετικές κυρώσεις. Στόχος είναι να έχουμε μια ομοιόμορφη εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε ανάλογα αποτελέσματα τα οποία θα πορέουν από τη σωστή αυστηρή επιβολή της Τελωνιακή Ένωσης. Να ευχαριστήσω την Κωνσταντ Λεγκρίπ και την Ευελίν Γκέπχαρτ για την ε, εργασία τους, για την έγκριση του σχεδίου ε, κανονισμού και είμαι απεπισμένος ότι και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να συνεχίσουν με την υποφασιστικότητα το έργο το οποίο είχε επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Αντώνιο Κορέα Ντεκάμπος για την πολύ αποτελεσματική εργασία του όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της καταπολέμησης της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της τροποποίησης του κανονισμού 515 κάθετος 97 για την αμοιβαία υποστήριξη. Βλέπω ότι ε, η έκθεση αυτή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινολεπτικής θητείας και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Μολονότι επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ στο ζήτημα των τελωνίων, υπήρξε και ένα δεύτερο κλάδο ο οποίο μα απασχόλησε ιδιαίτερα και αυτό έχει να κάνει με τη φορολογία. Ιδιαίτερα στα πλαίσια τη ολοκλήρωση τη ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα και για τον τομέα αυτό και όλο ιδιαίτερο για την φορολογία του ηλεκτρονικού εμπορίου και για το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά κάποιες τρέχουσε τρέχουσες πρωτοβουλίες. Την 1η Ιανουαρίου του 2015 θα έχουμε νέους κανόνες φόρου θέμενη αξίας για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις, επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές στο χώρο κατανάλωσης. Συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές και με τον εμπορικό κλάδο για να δημιουργήσουμε μια ενιαία θηρίδα εξυπηρέτησης One Stop Shop προκειμένου να επιτρέπουμε τελικά στους εμπόρους να μπορούν να καταχωρούνται και να, το, διαχειρίζονται το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλουν στις συναλλαγές που έχουν με καταναλωτές από άλλα κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τον Πάμπλο Αρία Σεκεβερία για την έκθεσή του όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο οποίο μα ζητεί να διευρύνουμε το πεδίο αυτού του one-stop shop και συμφωνώ μαζί του. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η νομοθεσία αφόρου προσθέμενη αξία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο και ιδίω όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε εξαιτία των εμποδίων αυτών αποθαρρύνονται από τον να διαστροποιούνται παγκοσμίω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βελτιώσουμε περισσότερο την πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίε MIDI έχουν ξεκινήσει μια προπαρασκευαστική εργασία, καθώ επίση και μια μελέτη αντικτύπου. Η εργασία αυτή θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει τι δέουσε αποφάσει. Τα επόμενα επίση χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει, θα πρέπει να βρει μάλλον λύσει για την φορολόγηση τη ψηφιακή οικονομία θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να φορολογήσουμε τους παράγοντες στην οικονομία, αυτή την ψηφιακή οικονομία, προκειμένου να έχουμε μια ισότιμη φορολογία, η οποία όμως δεν θα λειτουργεί, δεν θα αντιβαίνει στην ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη για το σημαντικό αυτό κλάδο δεν υπάρχουν πρόχειρε ή γρήγορε λύσει που θα μπορούσαν να βρεθούν στον τομέα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βασιστεί στα συμπεράσματα τη υψηλόβαθμη ομάδα εμπειρογνώμων για την φορολόγηση τη ψηφιακή οικονομία, συμπεράσματα τα οποία θα παρουσιαστούν το καλοκαίρι 2014. Κυρίε και κύριοι, ολοκληρώνω στο σημείο αυτό να σα ευχαριστήσω. Είμαι στη διάθεσή σα για παρατηρήσει και ερωτήσει και θα ήθελα να σα πω ότι ήταν πραγματική τιμή για μένα να συνεργαστώ μαζί σα. Σα ε, εύχομαι κάθε τύχη για το μέλλον, είτε, είτε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλο ιδιαίτερο τον άνθρωπο εκείνο που χάρη στην προσωπική του συμβουλή καταφέραμε να πετύχουμε καθοριστικά αποτελέσματα. Αναφέρομαι σε σένα, Μάλκομ. Η δική σου η προσωπική συμβολή και συμμετοχή συνέβαλε πάρα πολύ σε επιτυχίες της κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής. Αναφίβολα πιστεύω ότι ε, οι εξαιρετικέ σου ικανότητε ω πρόεδρο, η δυνατότητά σου να βρίσκει λύσει, η αποφασιστικότητά σου πραγματικά ήταν καθοριστικέ. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να σε ευχαριστήσουμε όλου ιδιαίτερω για την ε, εξαιρετική σου αυτή ηγεσία. Και λυπάμαι που βλέπω ότι δεν θα συνεχίσει το έργο σου. Πραγματικά έχει θέσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για οποιονδήποτε σε διαδεχθεί. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και προσβλέπω συζήτηση που θα ακολουθεί. Σα ευχαριστώ. Um, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τα πολύ γενναιόδωρα λόγια σας σε σχέση με μένα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι αναφέρατε ότι πολλά μέλη της Επιτροπής μας εργάστηκαν σκληρά στα εγχειρήματα αυτά, γιατί φυσικά παίζουν σημαντικό ρόλο για να είναι αποτελεσματική η Επιτροπή μας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ αποτελεσματικά τα μέλη αυτά και εγώ απλώς προσπάθησα να διευκολύνω το έργο αυτών των μελών για το τόσο αποτελεσματικό έργο της Επιτροπής μας. Μας είπατε ότι έχουμε επιτύχει πολλά και μας θυμήσατε και το έργο το οποίο έχουμε φέρει σε πέρας και το οποίο τώρα πια αρχίζει να εφαρμόζεται και αποδίδει καρπούς για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις που είναι και ο στόχος της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε περίπου μισή ώρα για συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις. Κύριε Στάλε, Σφάπ, ο κύριος Κουρία Ντεκάμπους, ο κύριος Μάντερς. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Κρόιτσμαν, μάλιστα, η κυρία Ρούλα. Κύριε Σφάπ, ναι, σας έχω καταγράψει. <clears throat> Κάποιος που δεν θέλει να λάβει το λόγο ίσως. Εντάξει. Λοιπόν, σε ομάδες των τριών, αν θέλετε, Ξεκινώ με την κυρία Στάιλερ, μετά ο κύριο Σφάμπ και ο καθηγητή Κουρέα Αντικάμψ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ ιδιαίτερα και εσά κύριε Πρόεδρε. Δύο σημεία που θέλω να αναφέρω. Το πρώτο για αυτό που είπατε για την ε, ε, ψηφιακή οικονομία και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Εγώ έχω ξεκινήσει μια ηλεκτρονική ε, εκστρατεία για να μπορέσουν να ενσωματωθούν τα βιβλία αυτά σε ψηφιακές αγορές ώστε να μην είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν χρήματα οι οποίοι μπορούν να υποφελούνται από τα ψηφιακά βιβλία. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα για το θέμα τη φορολογία αυτών των ηλεκτρονικών βιβλίων και τα άλλα συναφή θέματα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι το θέμα της φοροαποφυγής που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ των πολιτών μας. Στο δικό μου κράτος μέρο, υπολογίζουν ότι είναι από 15 έως 25 δισεκατομμύρια λίρε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν στα νοσοκομεία, στα σχολεία και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει και οι πολυεθνικές αλλά και τα πλούσια άτομα να συμβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σωστή φορολογία και πρέπει λοιπόν να αλλάξει η συμπεριφορά τους και να σταματήσει η φοροαποφυγή. Και εμείς χαιρόμαστε για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την καλή διακυβέρνηση αλλά βλέπω ότι υπάρχουν μονάχα δύο θέσεις οι οποίες δίνονται σε εργασιακές ενώσεις και μήκη όταν οι 15 άλλες δίδονται σε επιχειρήσεις. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη ισορροπίας. Πρέπει αυτός ο φορέας να δώσει πληροφορίες και αναφορές στο Κοινοβούλιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί η φοροαποφυγή και θα μπορεί να υπάρχει δίκαια φορολογία για όλους. Ευχαριστώ Κάθριν, ο Άνδρες Σφάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ Είχα ζητήσει προηγουμένως το λόγο, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να προσθέσω προηγουμένως τα λόγια μου. Ευχαριστίας για σας για το θαυμάσιο έργο σας και ελπίζω ότι και απόψε και σε άλλες ευκαιρίες ελπίζω ότι θα έχουμε περαιτέρω ευκαιρίες για να συζητήσουμε. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα όμως αυτά να τα καταγράψω στα πρακτικά και θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματος της ομάδας του ΕΛΚ τον Επίτροπο Σεμέτα για τα λόγια του. Και εγώ θέλω να προσθέσω λοιπόν τις δικέ μου ευχαριστίες και να αποτίσω φόρο τιμής όπως και οι άλλοι συνάδελφοι και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είμαστε απόλυτα απευθυσμένοι ότι έχουμε επιτύχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε κύριε Επίτροπε ότι οι πολίτες ενώπιον των ευρωπαϊκών εκλογών δεν ενδιαφέρονται μονάχα να βλέπουμε τα επιτευχθέντα, αλλά φυσικά ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτά τα οποία έχουν ακόμα παραμείνει αν, ανεκτέλεστα και αυτά πρέπει να γίνουν για το μέλλον. Και επειδή έχει ξεκινήσει ήδη και η προεκλογική εξατία θέλω να επανέλθω σε αυτά που είχαμε συζητήσει το 2009. Τότε αναφερθήκαμε στο τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε στη φορά η κυρία Στάιλερ και ιδίω για θέματα καπνικά, καπνικών προϊόντων, όπου έχουμε τον νέο αυτό κανονισμό. Παρ' όλα αυτά δεν επετέθησαν πολλά θέματα, όπως και στο παρελθόν και σήμερα τα κράτη-μέλη δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμα να μπορέσουν να έχουν ενιαία φορολογία των καπνικών προϊόντων σε όλη την ε, ε, Ευρώπη. Βασίζονται περισσότερο στη δυνατότητα να αντλούν περισσότερα φορολογικά έσοδα σε βάρος των άλλων. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε ένα ενίο καθεστώ θα ήταν καλύτερο για όλα τα κράτη-μέλη και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα για το μέλλον αυτή την πλευρά τη Κομισιόν. Θα ήθελα όμω να ακούσω τη δική σα άποψη για το τι μπορούμε να περιμένουμε εμεί ότι η επερχόμενη Κομισιόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει πιο έντονα. Και εδώ πιστεύω ότι οι φόροι οι οποίοι συνδέονται με συγκεκριμένα προϊόντα από τη δική μου πλευρά θα πρέπει να είναι πιο έντονοι και πιο καλά σταθμισμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχετε λοιπόν μια ατζέντα η οποία θα αλλάξει το μέλλον. Ο καθηγητή Κουρέα Ντεκάμπου. Και κλείνουμε τον πρώτο γύρο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα αγαπητέ κύριε Επίτροπε. Και εγώ θέλω να επαναλάβω φυσικά πιο σύντομα και από τους άλλους τις ευχαριστίες μας προς τον Μάλκομ και προς ε, εμάς. Θέλω να υπογραμμίσω την εξαιρετική διδακτική ικανότητα που είχε για τους βουλευτές που ήταν πιο, ήταν λιγότερο πεπειραμένοι για τα θέματα αυτά. Όταν ξεκινήσαμε το έργο της Επιτροπής μας, τότε ήταν της μόδας το σύνθημα κόπωση της εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει όμως αυτή την κόπωση τώρα και παρά το γεγονός ότι αυτή η διατύπωση δεν έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στο στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Σεμέτα. Νομίζω ότι χάρη στη βοήθεια και της δικής μας Επιτροπής μπορέσαμε να ξεπεράσουμε αυτή την υποτιθέμενη κόπωση της εσωτερικής αγοράς. Αλλά βλέποντας τους τρεις επιτρόπους που θα αντιμετωπίσουμε, που αντιμετωπίζουμε στους τομείς αρμοδιοτήτων μας, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη και ίσως αυτό είναι μονάχα το ορατό τμήμα του Παγοβούνου, αλλά Νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό ότι μπορέσατε και μεταξύ σας να κατανείμετε τις αρμοδιότητές σας με επιτυχή τρόπο σε έναν κόσμο που ήταν τόσο πολύπλοκος και λειτουργήσε αυτό πολύ καλά. Όλοι θα μπορούσαν να πιστεύουν καταρχήν ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει σωστό συντονισμό, αλλά εσεί πετύχατε να διαιρέσετε τι αρμοδιότητέ σα με αποτελεσματικό τρόπο. Εγώ παρέμεινα εντυπωσιασμένο με την τεράστια εργασία που έγινε στον τελωνιακό τομέα. Πριν από 30 χρόνια ποιος θα φανταζότανε ότι με την εξάλληψη των εθνικών τελωνίων μεταξύ των χωρών μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα επίτροπο του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων έχει να κάνει με τη ρύθμιση των τελωνιακών θεμάτων. Αυτό είναι, θα έλεγα, και αποτέλεσμα της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των οικονομικών σχέσεων και της πολυμορφίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον παγκόσμιο κόσμο του εμπορίου ιδίως. Για το μέλλον. Είναι σημαντικό ότι ούτε εγώ προσωπικά ούτε ο Επίτροπος ε, Σεμέτα θα παραμείνουν σε αυτό το χώρο για τα τελωνιακά θέματα και την ενιαία αγορά. Αυτά τα οποία λέω λοιπόν δεν έχουν πραγματικά ένα ε, αποδέκτη ούτε καν τον ε, Μάλκομ για, τις επόμενες, ε, για την επόμενη επιτροπή και τους επόμενους κοινοβουλευτικούς. Θέλω όμως να τονίσω τα εξή θέματα για το ψηφιακό εμπόριο. Καταρχήν νομίζω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα έχει μεγάλη και ραγδαία ανάπτυξη ο τομέα λοιπόν του ψηφιακού εμπορίου, οπότε θα πρέπει να μα απασχολήσει ιδιαίτερα. Δεύτερον, το θέμα τη εναρμόνιση του ΦΠΑ. Εγώ δεν είμαι τόσο φιλόδοξος ώστε να πιστεύω ότι στα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορέσουμε μια πλήρη, να φτάσουμε σε μια πλήρη δημοσιονομική εναρμόνιση ό,τι αφορά τους καταναλωτικούς φόρους και το ΦΠΑ. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις ανάγκες και να ρονταριζόμαστε στα επόμενα πέντε χρόνια. Και πιστεύω επίσης ότι η εναρμόνιση της εμπορικής νομοθεσίας μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα και εδώ είμαι αισιοδόξο γιατί έχουμε κάνει μερικά σημαντικά βήματα προ την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι και εμεί και η νομική επιτροπή μαζί μα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για το μέλλον ότι θα αποκομίσουμε κάποια θετικά αποτελέσματα στην επίτευξη μεγαλύτερη εναρμόνιση για την εμπορική νομοθεσία. Αυτά λοιπόν για να πω ότι το έργο τη Επιτροπής μα τα τελευταία πέντε χρόνια δεν ήταν ε, μονάχα το κομμάτι το οποίο σήμερα είναι ορατό, αλλά ήταν και ένα έργο το οποίο σε μεγάλο βαθμό υπόγεια ή αόρατα θα κρατήσει την αξία του για το μέλλον και θα μπορέσει να είναι η βάση της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ημών και της ε, επερχόμενης Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ τώρα να ζητήσω από τον Επίτροπο Σεμέτα να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και θα ακολουθήσει μια ομάδα πάλι τριών ή τεσσάρων βουλευτών. Ευχαριστώ. Νιώθω σαν να είμαι στην Επιτροπή οικονομικών ε, θεμάτων. Έχω να αντιμετωπίσω θέματα τα οποία βέβαια είναι πολύ σημαντικά τα φορολογικά θέματα και για τη δική σας ε, επιτροπή και σε όλη αυτή τη διάρκεια της θητείας μπορέσαμε να βάλουμε ψηλά τον πύχη και την ατζέντα που έχει να κάνει με τα θέματα αυτά τα φορολογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ότι υπάρχει πάντα αμύωτο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά για την ψηφιακή τώρα οικονομία και ιδίω για τη μεταχείριση των, φορολογική μεταχείριση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Όπως είπα στην αρχή μου, στην αρχική μου παρέμβαση, έχουμε μια ομάδα υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων, η οποία επεξεργάζεται συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ψηφιακή οικονομία, είτε σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της ψηφιακής οικονομίας, αλλά επίσης και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτό της φοροαποφύγης το οποίο επισημάνατε. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πραγματικά σοβαρά προβλήματα. Η έκθεση λοιπόν αυτής της ομάδος ε, εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου πιστεύω ότι θα μπορέσει να δημοσιευτεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και προσβλέπω και εγώ στο να δω, να δω αυτές τις συστάσεις Σε ό,τι αφορά τώρα τα ποσοστά του συντελεστέ, ΦΠΑ, η Κομισιόν ε, έχει μια έκθεση αντικτύπου και βάσει αυτής αξιολογεί τον αντίκτυπο της μείωσης συντελεστών ΦΠΑ επί τη βάση μιας σειράς κριτήριων και επί τη βάση αυτής της αξιολόγησης και φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Επιτροπή σας είναι ιδιαίτερα προσιλωμένη στο να παρακολουθεί και αυτές τις αξιολογήσεις. Πρωτού όμως καταλήξουμε σε τελική απόφαση θα πρέπει να γίνει αυτή η ενδελεχής αξιολόγηση για τα θετικά και αρνητικά στοιχεία μιας οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και ενέργειας της Κομισιόν. Όλα αυτά λοιπόν συνεχίζονται ακόμα και προσπαθούμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα στοιχεία ώστε η τελική μας αξιολόγηση να μπορεί να δημοσιευτεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας. Για τα θέματα φοροαποφυγής τώρα. Υπάρχουν πολλά, πολλές ενέργειες οι οποίες είναι εξελίξει στον τομέα αυτό. Ξεκινώ με τα σχέδια δράσης μας για το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και τι συναφείς ε, συστάσεις που έχουν απευθυνθεί στα κράτη-μέλη για την εισαγωγή ενό γενικού κανόνα κατά τη καταχρηστικής συμπεριφοράς στα φορολογικά θέματα και άλλων σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν και την ε, δημιουργία μιας πλατφόρμας όπως ελέγχθη για την καλή διακυβέρνηση στα φορολογικά. Ξέρω ότι υπήρξαν κάποιες επικρίσεις για την σύνθεση αυτής της πλατφόρμας αλλά οι υπηρεσίε μου με διαβεβαίωσαν ότι αυτή η επιλογή έχει γίνει επί αντικειμενικής βάσεως και αυτό το έργο το οποίο έχει πρακτικό χαρακτήρα δεν θα επηρεαστεί από δυνητικές ε, κατά κάποιο τρόπο ελλείψεις ισορροπίας σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των μελών της πλατφόρμας και εξάλλου οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ήταν παρούσες σε αυτή την πλατφόρμα ήταν ιδιαίτερα ενεργές στο να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και με τον τρόπο αυτό έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στο έργο της δημιουργία αυτής της πλατφόρμας χρηστής διακυβέρνησης. Προσβλέπω λοιπόν στο να εδρεωθεί ο ρόλος αυτής της πλατφόρμας ως η ομάδα η οποία θα μπορέσει να παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων οι οποίε προβλέπονται από το σχέδιο δράση τη Κομισιόν και έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα του πώς τα κρατημέλη αντιμετωπίζουν αυτές τις γενικές αρχές κατά της καταχρηστικής συμπεριφοράς και έχουμε εξάλλου πρόθεση να συζητήσουμε το θέμα του πώς θα εφαρμοστούν οι συστάσεις για τον αγώνα κατά των φορολογικών παραδείσων Γενικά λοιπόν το έργο αυτής της ομάδας είναι ιδιαίτερα θετικό και με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι απαντώ στο ερώτημά σας πρέπει να προχωρήσουμε και με προτάσεις ιδεών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και αυτό μπορεί να είναι και ένα έναυσμα για μελλοντικέ νομοθετικές προτάσεις από την πλευρά της Κομισιόν για τα καπνικά προϊόντα και τη φορολογία τους. και εγώ συμφωνώ ότι το θέμα της λαθεμπορίας τσιγάρων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπολογίζουμε ότι, υπάρχει μια απώλεια περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κάθε χρόνο λόγω του λαθεμπορίου τσιγάρων. Γι' αυτό πέρσι υιοθετήσαμε μια στρατηγική, μια πλήρη στρατηγική αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας τσιγάρων. Και αυτή η στρατηγική επικυρώθηκε από το Συμβούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτού του έργου, το λεγόμενο πρωτόκολλο FCTC για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε αυτό το πρωτόκολλο. Η Κομισιόν συγκεκριμένα υπέγραψε αυτό το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το οποίο είναι σημαντικό σήμερα είναι να μπορέσουμε να ακυρώσουμε αυτό το πρωτόκολλο και να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε. Γιατί μας δίνει πολύ καλύτερες δυνατότητες αυτό το, το πρωτόκολλο για την ανείχνευση και παρακολούθηση των παρτίδων σιγαρέτων πέραν αυτού που προβλέπεται στην αρμόδια οδηγία. Το FCDC επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητος σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη, τον πλανήτη μας και είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου σε όλο τον κόσμο και ιδίω στα μεγαλύτερα κέντρα κατανάλωσης όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα κτλ. από τα οποία έρχονται πάρα πολλά ε, προϊόντα λαθρεμπορίας. Για το φόρο κατανάλωσης ε, για τα καπνικά προϊόντα προβλέπουμε επίσης να διατυπώσουμε προτάσεις για την τροποποίηση των οδηγιών που διέπουν αυτά τα προϊόντα με στόχο να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Για τους συντελεστές λοιπόν υπάρχουν συμφωνίες για μια μεταβατική περίοδο. Αυτό είναι μια συμφωνία που είναι πριν από μερικά χρόνια και για πολλά κράτη-μέλη μόνο μετά από το 2018 εκπνέουν αυτές οι μεταβατικές περίοδοι. Θα χρειαστούμε επομένω λίγο περισσότερο χρόνο για να δούμε πώς το νέο σύστημα φορολογικών συντελεστών θα λειτουργήσει στην πράξη. Υπάρχουν όμως και άλλες ελλείψεις στην οδηγία για τα καπνικά προϊόντα που θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε με την ευκαιρία αυτή. Και τώρα ανέλθω στα σχόλια του καθηγητού Κουρέα Ντουκάμπους. Σύμφωνο ότι είναι πολύπλοκο το χαρτοφυλάκιό μου και υπάρχει πολλή επεξεργασία πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερα τεχνικά θέματα όπου είναι απαραίτητη η εμπειρογνωμοσύνη. Ελπίζω όμως ότι με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας και με τη βοήθεια και των κρατών μελών έχουμε επιτύχει πολλά κατά τη διάρκεια της ε, τρέχουσας θητείας και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ευγνώμων για το πολύ καλό έργο που έγινε με τον τελωνιακό κώδικα, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να πιστεύει, όπως πήγε ο καθηγητής Ζεκάμπους, ότι ένα τόσο πολύπλοκο έγγραφο θα μπορούσε να εγκριθεί σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα τα θέματα αυτά και ο κανονισμός για την εφαρμογή του κώδικα δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για την εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα. Δεν πρόκειται τώρα να διεξέλθω όλα τα στοιχεία της πρότασης, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα στάδιο όπου σε νομοθετικό τουλάχιστον επίπεδο έχουμε στα χέρια μας ένα σύστημα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης. Θα πρέπει εδώ να επενδύσουμε και στα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης του, του συστήματος αυτού και ανέφερα ήδη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ε, θητείας θα έρθουμε με ένα σχέδιο για την ε, διακυβέρνηση, τη μορφή αυτής της διακυβέρνησης και το επερχόμενο κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις ιδέες και επίσης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διαχείριση του κινδύνου. Θέλουμε να βελτιώσουμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του κινδύνου για να είναι πιο στοχευμένη η αντιμετώπιση και να έχει και ένα πιο εγκάσιο χαρακτήρα, ώστε με τον τρόπο αυτό να υπάρχει δυνατότητα να συμμεριζόμαστε πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών και να χρησιμοποιούμε ενιαία συστήματα διαχείρισης κινδύνου. Αν μπορέσει λοιπόν αυτή η ρύθμιση να εφαρμοστεί και να εφαρμοστεί θετικά, θα επιτρέψει και στα κρατημέλη να εξοικονομήσουν σημαντικά κονδύλια σε ό,τι αφορά το κόστος των τελειωνιακών ελέγχων και φυσικά και οι εμπορευόμενοι θα εξοικονομήσουν πολλά χρήματα γιατί θα υπάρχει αντιμετώπιση τους μόνο επί τη βάση του προφίλ κινδύνου και όχι με σποραδικό ή αποσπασματικό τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν, να συνεχιστεί η προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και πιστεύω ότι θα χρειαστούμε να βασιστούμε σε όλα αυτά που έχουν γίνει στον χώρο αυτό σε διεθνές επίπεδο μετά από την έγκριση της ε, Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου σε επίπεδο ΠΟΕ πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι φυσικά προς το δικό μας ε, συμφέρον να εφαρμοστεί πλήρως αυτή η συμφωνία δεδομένου ότι είμαστε η εμπορική οντότητα η οποία είναι πιο ενεργή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οικονομική μας ανάπτυξη και ευμάρεια λοιπόν εξαρτάται ιδιαίτερα από την ορθή λειτουργία του εμπορίου, γι' αυτό μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν προς την βελτίωση των καταστάσεων και να άρουμε τα εμπόδια τα οποία εμποδίσουν τις εμπορικές συναλλαγές. Πέρα λοιπόν αυτών τα οποία αναφέρατε εσείς ως δυνητικές προτεραιότητες, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε και την προσοχή μας και στον διεθνή χώρο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου στο, στα πλαίσια του ΠΟΕ και αυτό θα είναι το σημαντικό εγχείρημα για την επερχόμενη επιτροπή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγο ακόμη χρόνο για κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να είστε σύντομοι. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε να πάτε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών. Μάντες, Κρόιτσμαν, Ρούλε, όχι, όχι Ρούλε. Και η κυρία Λάγκεν. Θέλει κανεί άλλο το λόγο? Ωραία. Κύριε Μάντερς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτροπε για τις απαντήσεις σας όσον αφορά τη φορολόγηση και τους φόρους κατανάλωσης. Ε, και την ε, ψηφιακή αγοριά, αγορά. Πολλές ε, φορές ε, μου έχουν, με έχουν πάρει επιγόντως τηλέφωνο γιατί πάρα πολλές ε, ε, υπηρεσίες δεν μπορούν πια να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, καταλαβαίνω όμως ότι και εσείς χρειάζεστε χρόνο για να ολοκληρώσετε τη δουλειά σας. Καταλαβαίνετε ότι η ψηφιακή αγορά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Ελπίζω να μην χρειαστούμε λοιπόν δύο χρόνια για μια πολύ καλή μελέτη και τα πορίσματα αυτής, γιατί τότε μπορεί να, να έχουμε καθυστερήσει πολύ σε σχέση με αυτά που είπε ο Ανδρέας Σφάμπ. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μάχη ε, για το πετρέλαιο ε, στις ε, σε μερικές χώρες μεταξύ των οποίων και τη δική μου χώρα. Η Ολλανδική κυβέρνηση αύξησε δραματικά τον ειδικό φορό κατανάλωσης και ξέρετε ότι αυτό βέβαια είναι ξέρετε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς μπορούν οι Ολλανδοί Ολλανδοί να πάνε στο Βέλγιο να κάνουν τα ψώνια τους, ειδικότερα στις μεθοριακές περιοχές ε, και βλέπουμε τώρα, κυρίως σε περιοχές αυτές, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση ε, τζίρου και νομίζω ότι τελικά ε, δημιουργείται ένα ε, πεδίο που δεν είναι καθόλου ισότιμο. Ε, ίσως θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μια παρέκκληση από τον κανονισμό για την ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη γιατί πραγματικά είναι επίγον για τους ανθρώπους αυτούς και θα ήθελα πραγματικά να ε, σας κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Όσον αφορά τώρα τις ψηφιακές ε, εφημερίδες και εκείνες ε, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για τη δουλειά σας. Πολλές φορές έχετε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ε, ιδιοκτησίας από τα τελωνία. Αλλά αυτά που έχω εγώ διαπιστώσει είναι ότι οι τελωνιακές αρχές δεν ε, είναι ε, σε ισότιμη θέση σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε μερικά κράτη-μέλη πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν για τα τεολονία και υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη όπου είναι πολύ ολιγάριθμο το εργατικό δυναμικό. Δεν ξέρω βέβαια αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επιβάλλει τον αριθμό των εργαζομένων στις τελωνιακές αρχές. Μήπως θα μπορούσαμε όμως να έχουμε μια καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, γιατί όταν υπάρχει ένας κανονισμός ε, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών ε, και δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι για να γίνει σωστά η καταπολέμηση ε, της απάτης και η προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών, δεν θα δουλέψει ο κανονισμός ε, αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος και η κυρία Κορίν Λάγκεν. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να έρθω σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα της, ε, του άκτους της γραφειοκρατίας, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλο και πιο επίκαιρο είναι αυτό το θέμα για πράγματα τα οποία είναι συγκρίσιμα και παρόμοια. Πολλές φορές υπάρχει αντιμετώπιση πολύ διαφορετική ώστε να υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση για ορισμένου. Υπάρχουν διαφορετικές ε, χάρη ρυθμίσεις για προϊόντα τα οποία περνούν από το τελωνίο και άλλα τα οποία δεν περνούν. Έχουμε στην Χέση διάφορες διαδικασίες πιστοποίησης οι οποίες κοστίζουν 25 ε, χιλιάδες ευρώ και 300 ώρες για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα θέμα όπου τίθεται να αμφιβόλο η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί λένε ότι οι επιχειρήσεις ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας τρόπος να είναι πιο εύκαμπτη η γραφειοκρατία. Βέβαια λοιπόν γενικά το θέμα αυτό της ίσης μεταχείρισης των επιχειρήσεων και της μείωσης γενικά του γραφειοκρατικού άκτους. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Να δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει και να μας, πει και κάποια, να μας κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Σε σχέση με τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Μάντερς, χαίρομαι ιδιαίτερα που θέλετε να μου δώσετε τόσο πολύ σημαντικές εξουσίες στον τομέα της ε, φορολογίας, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν ε, μου δίνουν τέτοια, τέτοιες εξουσίες. Όλα τα φορολογικά ζητήματα που ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ρυθμίζονται από ε, το δίκαιο. Όταν ανεφέρθηκα στην ψηφιακή οικονομία, δεν είναι μόνο η ψηφιακή οικονομία, ε, υπάρχουν και αλλού μειωμένοι συντελεστές και η δική μου πρόθεση είναι πριν από το τέλος της θητείας να ολοκληρώσω τη δουλειά μου από αυτού και επί τη βάση της δουλειάς αυτής ε, θα υπάρξουν ενδεχομένως ε, μεταγενέστερες δράσεις. Αλλά δεν έχω φτάσει ακόμη στην παρέκκληση στην οποία αναφερθήκατε, δηλαδή στην παρέκκληση από την εφαρμογή ε, των, ε, της νομοθεσίας. Υπάρχουν κάποια ελάχιστα επίπεδα συντελεστών ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν τους δικούς τους φορολογικούς συντελεστές. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο υπάρχει συζήτηση για την, για τις, για την τροποποίηση της οδηγίας της φορολόγησης της ενέργειας. Ε, εξετάζονται τα ξεχωριστά συστήματα των κρατών μελών, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο τομέας και υπάρχει βέβαια και το θέμα της ε, ομοφωνίας. Πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση δεν βλέπω λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να λάβουμε αποφάσεις τάχιστα. τα κράτη-μέλη σέβονται τους ελάχιστους συντελεστές. Έχουμε ελάχιστους συντελεστές που πρέπει να την χάνουν σεβασμού και τα κράτη-μέλη έχουν κάποιες μεταβατικές περιόδους ε, μεν, αλλά έφτασαν ε, στο τέλος τους αυτές οι μεταβατικές περιόδους. Όταν μιλήσατε ας πούμε για το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία ή άλλα κράτη-μέλη, όλα αυτά τα κράτη ε, σέβονται τα ελάχιστα επίπεδα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε το τι κάνουν. Ίσως στο μέλλον να γίνει μια συζήτηση για το επίπεδο των ελάχιστων συντελεστών. Είναι μια συζήτηση που γίνεται στο Συμβούλιο στο πλαίσιο της ε, οδηγίας για την ε, φορολόγηση της ενέργειας. Τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολες αυτές οι συζητήσεις. Όσον αφορά το θέμα που έθεσε ο κύριος Κρόιτσμαν και την ε, ισότιμη, την, ίση εφαρμογή ε, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τις τελωνιακές αρχές είναι ένα από τα θέματα που ετέθησαν ε, και από τους επικεφαλείς των τελωνιακών αρχών των κρατών μελών και είναι ένα θέμα το οποίο θα θέλουμε, θέλουμε να αποτελέσει το επίκεντρο του οδηγού μας ε, για την εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα, γιατί το όραμά μου εμένα είναι ε, τα τελωνία σε όλα τα κράτη-μέλη να είναι περίπου ίδια. Η διαχείριση είναι βέβαια εθνική, αλλά θα έπρεπε να είναι κάτι σαν υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας, για να το πω έτσι. Αν πάει κανείς, ας πούμε, στη BNP Paribas, ε, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα πάει, είναι το ίδιο το σύστημα. Πρέπει λοιπόν μακροπρόθεσμα να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι παρόμοιο και στον τομέα των τελωνίων. Βέβαια, η ανταλλαγή των πρακτικών είναι πολύ σημαντική και εγώ ε, έγραψα στα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν ε, στις προτεραιότητες τους ε, στο πρόγραμμα, ε, στα διευθυντικά προγράμματα ε, να συμπεριλάβουν και τα τελωνία ως προτεραιότητα. Ίσως τα διαρθρωτικά ταμεία να μπορούσαν να βοηθήσουν ειδικότερα τις ανατολικές μεθοριακές περιοχές. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως μαζί σας ότι πρέπει να προσπαθήσουμε σε κάθε κράτος μέλος ε, τα, οι τελωνιακές αρχές να δουλεύουν στο ίδιο επίπεδο. Όσον αφορά τώρα την ε, απλοποίηση, αυτή τη στιγμή εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τις περισσότερες ε, προτάσεις ε, όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική τιμολόγηση 18 δισεκατομμύρια εξοικονόμηση θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για επιχειρήσεις, όπως επίσης και για τη δήλωση του ΦΠΑ. Του ΦΠΑ. είναι πολύ σημαντική ε, η νομοθεσία αυτή, γιατί 15 δισεκατομμύρια θα, μπορούσαμε να, θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν οι επιχειρήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι διαπραγματεύσεις για τον ε, τελωνιακό κώδικα της Ένωσης νομίζω ότι μας επέτρεψαν έναν ε, αποδεκτό συμβιβασμό για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να απλοποιήσουμε περισσότερο τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το σύστημα, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μερικές φορές τα κράτη-μέλη υπερθεματίζουν μερικές φορές ε, από νομοθετικής απόψεως, ε, δημιουργούν δηλαδή περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσπαθούμε βεβαίως να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Όμως το σύστημα αυτό των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων θα μπορούσε νομίζω να διευκολύνει τις ε, συναλλαγές ε, με έμπιστους ε, εμπόρους και όπου υπάρχουν εμπόδια πρέπει βεβαίως να αρθούν. Α, και κάτι ακόμη, μια και πρέπει να ολοκληρώσω τώρα την παρέμβασή μου. Θα θέλα μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής για την εξαιρετική συνεργασία Καταφέραμε πολλά στον τομέα αυτόν, που είναι πολύ τεχνικός, ειδικότερα στον πολύ τεχνικό τομέα των τελωνίων, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας στα τελωνία και είναι πολύ ε, σημαντικό να ε, βλέπουμε ότι τα τελωνία λειτουργούν σωστά. Αν υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα, αμέσως ε, θα έβλεπε κανείς τη σημασία των τελωνίων για την ε, ενιαία αγορά. Νομίζω ότι κάναμε πολύ μεγάλη πρόοδο κατά τη διάρκεια της θετίας αυτής. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους. Μάλκολμ, εσένα ως πρόεδρο όλος ιδιαίτερος να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία και την ε, αμοιβαία κατανόηση, την ε, δυνατότητα σε συμβιβασμών, ε, μερικές φορές σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Κύριε Επίτροπε, και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω πολύ θερμά εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής μας, εξ ονόματος των παρευρισκομένων και όλων των υπολείπων που δεν μπορούν να είναι σήμερα εδώ, αλλά που εργάστηκαν για τα ζητήματα των δικών σας αρμοδιοτήτων. Αρμοδιότητες τις οποίες όντως σημειώσαμε πολύ σημαντική πρόοδο, απομένουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να επιτευχθούν όπως το είπατε, αλλά ιδιαίτερα ο εξυγχρονισμένος τελωνιακός κώδικας, αλλά και άλλα σημαντικά μέτρα όπως η, αυτά τα οποία προβλέπονται στην έκθεση Κρόιτσμαν, το πρόγραμμα Τελωνία 2020, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ζήτημα το οποίο επεξεργαστήκαμε μαζί με εσά και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά, ο εγκεκριμένο οικονομικό φορέα, ζήτημα το οποίο πρέπει να σα απασχολήσει πολύ και στο μέλλον, προκειμένου πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι το νέο αυτό μέσο θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς. Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν σημαντικότατα επιτεύγματα και καταφέραμε πραγματικά πολύ επικοδομητικά να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσωπική σας συμμετοχή, για την αφοσίωσή σας αυτή που πραγματικά καθόρισε την ευτυχή έκβαση όλων αυτών των προτάσεων. Και να ευχαριστήσω προφανώς και τις υπηρεσίες σας και τους συνεργάτες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σας εδώ σήμερα και σας ευχόμαστε καλή τύχη σε οτιδήποτε κάνετε και εσείς στο μέλλον, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ουδής το γνωρίζει. Σας ευχαριστούμε πάντως ε, πολύ για το ότι καθοδηγήσετε πάρα πολύ καλά όλο αυτό το σημαντικό το χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστούμε. Okay. Uh, uh, Μάλιστα. Προχωράμε τώρα στα δύο επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Όσοι αποσιάζατε σήμερα το πρωί, ενδεχομένως να μην έχετε δει το email το οποίο σας έστειλα. Ο Επίτροπος Μιμίτσα δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει σήμερα το απόγευμα να μας μιλήσει. Ξέρω ότι έχει απογοητευτεί και ο ίδιος πάρα πολύ με αυτό έχει μια πολύ σημαντική έκθεση την οποία θα ήθελε να μας παρουσιάσει και ελπίζω ότι έχετε και εσείς αντίγραφα της έκθεσης αυτής. Λογικά όλοι σας πρέπει να έχετε αυτή την έκθεση, τη βλέπετε. Έχει να κάνει με την πολιτική για τους καταναλωτές. Σας προτείνω τώρα να εγκρίνουμε τις επιστολές για τον προπολογισμό θα δώσω σε λίγο το λόγο στον καθηγητή Κορέα Ντεκάμπος. Με απλή ψηφοφορία μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν πρόκειται για νομοθετική πρόταση. Δεν χρειάζεται λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία. Το μικροφόνο η παρέμβαση. Έχετε τις κάρτες σας ψηφοφορίες μαζί ή θα πρέπει... Πώς έχετε τις κάρτες σας. Για σηκώστε χέρι παρακαλώ. Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, θα κάνουμε έναν έλεγχο λίγο αργότερα. Και εγώ νομίζω ότι έχω την κάρτα μου. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία να σας πω ότι η διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου όσον αφορά την εργασία μας και μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής να αναφερθώ λίγο στα σημαντικότερα σημεία της δήλωσης αυτής. Θεωρώ ότι το μήνυμα είναι πολύ θετικό. Αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι ε, μάλλον συγχαίρει καταρχάς την ε, δική μας την Επιτροπή γιατί έθεσε πραγματικά τους καταναλωτές ε, στην καρδιά των εργασιών που κάνουμε γιατί προσπαθούμε πραγματικά να προστατεύσουμε τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό και προσπαθώντας να θεσπίσουμε από κοινού μία ατζέντα για την πολιτική καταναλωτών, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, μια καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, μια καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας πανευρωπαϊκά και έχουμε μια συνεχή προσαρμογή της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών στα νέα δεδομένα τα οποία συνεχώς εξελίσσονται. Όσον αφορά την εφαρμογή της ατζέντα για τους καταναλωτές, αυτή ε, δημοσιεύτηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η έκθεση ουσιαστικά την οποία έχετε μπροστά σας και ουσιαστικά μας υπενθυμίζει την εργασία που τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επιτελέσει για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και αποτελεί μια εξαιρετική βάση για την διευθέτηση κάποιων προβλημάτων που ακόμα εκκρεμούν όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών. Το γεγονός ότι θα πρέπει να επιβάλλει την νομοθεσία καλύτερα, το ότι θα πρέπει να διευθετήσουμε καλύτερα το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει το νέο ηλεκτρονικό ψηφιακό περιβάλλον το οποίο αναδύεται όλο και περισσότερο. Αυτά ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας διαβάσω την δήλωση αυτή και θα στείλω και στον Επίτροπο Μίμητσα ένα μήνυμα από τη δική σας την πλευρά και θα του πούμε ότι τον ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή την οποία μας προώθησε, που μας διαβίβασε, μόλον ότι δεν μπόρεσε βέβαια να είναι σήμερα εδώ πέρα μαζί μας για να μας μιλήσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Προχωράμε τώρα στο επόμενο σημείο της της διάταξης, έγκριση δύο επιστολών για τις προτεραιότητες για το προπολογισμό 2015, καθώς επίσης και κάποιες προτάσεις για πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κορέα Ντεκάμπος για να μας μιλήσει για τις επιστολές αυτές. Μπορείτε να πάρετε και υπόλοιποι το λόγο εφόσον το επιθυμείτε και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε για τις δύο αυτές επιστολές. Δεν υπάρχουν τροπολογίες, επομένως θα έχουμε μια και μοναδική ψηφοφορία για αυτές τις δύο επιστολές. Κύριε Καθηγητή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, το κείμενο το οποίο έχουμε στείλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ως γνωμοδότηση εξηγεί τις εγκάρσεις ενασχολήσεις μας και ανησυχίες μας. Υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά είναι ένα κομβικό τομέα για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά σχέδια, οι προτεραιότητές μας είναι το φόρουμ της ενιαίας αγοράς, που είναι μια αίτηση της ε, Επιτροπής μας ήδη από την αρχή τη τρέχουσας θητείας και για το σχέδιο Europe Travel, μια εφαρμογή για κινητά, για κινητές συσκευές, δηλαδή μια εφαρμογή που αφορά τα κινητά τηλέφωνα και τις ταμπλέτες όπου περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίε υποστήριξης προς τους ε, ταξιδεύοντες. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γραμματεία της Επιτροπής μας και φυσικά και τους σκιώδεις εισηγητές για την έγκριση αυτής της ε, σύστασης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Έχετε το κείμενο της επιστολής στο παράρτημα της έκθεσης που απεστάλλει και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ε, υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα, όλους τους συναδέλφους και ιδίω για τις πάρα πολύ χρήσιμες τροπολογίες, χάρη στις οποίες το κείμενο και η επιστολή έχουν εμπλουτιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Θέλει καμία άλλη πολιτική ομάδα να πάρει το λόγο. Ωραία, οπότε να ψηφίσουμε. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Όποιοι δεν έχουν τις κάρτες του σηκώστε το χέρι. Δύο επιστολές. Η πρώτη επιστολή είναι προτεραιότητε ΣΥΜΚΟ για τον προϋπολογισμό 2015. Υπέρ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. We have okay. All right, anyone can put their card in. Ψηφίσατε όλοι. 18 υπέρ, καμία ψήφος ε, κατά και καμία αποχή. Πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία για την ε, πρόταση των προπαρασκευαστικών πράξεων και των πιλωτικών προγραμμάτων έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 18 ψήφοι υπέρ, ε, καμία ψήφος κατά και καμία αποχή. θα συμπεριλήφθουν οι επιστολές αυτές στις προτάσεις μας για τον προϋπολογισμό του 2015. Θα τις ε, μεταφέρουμε στον εισηγητή μας. 10, 5 παρα 10 αναμένουμε τον κύριο Μπαρνιέ. Στη χώρα μου είναι η κατάλληλη στιγμή για να πιούμε τσάι. Οπότε διάλειμμα για τσάι. πέντε η ώρα ή και λίγο νωρίτερα, παρακαλώ να είστε εδώ, για να είμαστε εδώ γέρος για τον κύριο Μπαρνιέ. Μετά από την παρέμβαση και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του κυρίου Μπαρνιέ θα υπάρξει κοκτέιλ απ' έξω από την αίθουσα. Έρχονται όμως τώρα επισκέπτες της κυρίας Βάιλερ. Έρχονται δυστυχώς σε λάθος ώρα. Ευχαρίστω να τους ε, μιλήσω όμως ε, έξω από την αίθουσα αν θέλουν. just welcome to talk to. Okay. Barbara, did you want to just... Barbara, θέλεις να εξηγήσεις ε, στους επισκέπτες σου ότι έχουμε διάλειμμα. Use the microphone if you like. You can... Με το μικρόφωνο αν θέλεις. Με το μικρόφωνο. Geht das? Ja. Ja, wunderbar. Dann würde ich meine Gruppe bitten, mal die Kopfhörer aufzusetzen. Για τους ελληνόφωνες καλεσμένους της κυρίας Βάιλερ. Θα αναλάβει ο πρόεδρος να σας εξηγήσει. Sorry. English? Yeah, German? Uh, channel number one is German, yes. Uh, so can I, um, uh, can I, as chairman of the committee, warmly welcome you to uh, the European Parliament. A visit to Mrs. Weiler, who is a very hard-working and respected member of our committee. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Βάιλερ, η βουλευτή σας είναι ένα από τα πιο σκληρά εργαζόμενα μέλη αυτής της Επιτροπής. Δυστυχώς ο Επίτροπος κ. Μίμητσα, ο οποίος ήταν να μας επισκεφθεί τώρα, έχει αρρωστήσει και δεν θα έρθει στην συνεδρίασή μας. Γι' αυτό τον καιρό Γι' αυτό το λόγο μάλλον εγώ έχω αναγκαστεί να διακόψω τη συνεδρίαση της Επιτροπής κάτι το οποίο συμπίπτει με την Βρετανική παράδοση για τεϊοληψία και θα επανέλθουμε στις 5 με τον κύριο Μπαρνιά. Είναι κάτι το οποίο ήταν απρόπτο και εξεφεύγει από τις δυνατότητες ελέγχου μας. Αν θέλετε λοιπόν μπορώ να σας συναντήσω έξω ή αν θέλετε να απαντήσω κάποιο ερώτημα της κυρίας Βάιλερ ή ημών με Y και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάλκον Χάρμπορ είναι από το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα αλλά παρόλα αυτά είναι υποστηρικτής της Ευρώπης και υποστηρικτής της ε, ενιαίας αγοράς και γι' αυτό έχει υποστηριχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια και από την Επιτροπή μας και ακούσατε θα, θα έρθει αργότερα ο Επίτροπος Μπαρνιέ ε, κανονικά θα είχαμε πάντα τη δυνατότητα να ακούσετε εδώ την, ε, τι συμβαίνει στη συνεδρίαση, αλλά φοβάμαι ότι επειδή αυτό ήταν απρόπτο, θα πρέπει να σας... Ε, δεν μπορούμε να ακούσουμε. Εδώ πέρα, αν δείτε εδώ πέρα πώς είναι η αίθουσα, βλέπετε ότι στα δεξιά είναι η φιλελεύθερη και η συντηρητικοί και αριστερά είναι οι σοσιαλιστές. Οι διερμηνείς είναι πάρα πολύ στενοχωρημένοι για αυτή τη διακοπή της συνεδρίασης που ζήτησε ο κύριος Χάρμπορ. Δίπλα στον Μάλκον Χάρμπορ είναι ο Πάρος Κωνσταντόπουλος από την Ελλάδα, ο, ο οποίος είναι Έλληνας αλλά καταλαβαίνει γερμανικά και δίπλα του είναι ο Μητροφάνης Ρέπο, ένας σοσιαλιστής από τη Φιλανδία, ο οποίος είναι τελείως αξιόλογος. Λοιπόν, μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην διακοπή ΤΕΙΟΥ. Έτσι. Γίνεται με τις ε, συνεδριάσεις. Δεν ξέρω τώρα αν προβλέπετε να χτιστούν και άλλες καμπίνες ε, διερμηνέων να έρθουν και άλλες χώρες μέλη. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει και πολλής χώρος που έχει μείνει. Έχουμε πολλές καμπίνες σήμερα. Έχουμε και κροατική διερμηνία. Γιατί ο κύριος Μίμητσα θα μιλούσε στα κροατικά. Είναι πάντα καλόδεκτη. Σας λέω και πάλι λοιπόν ότι θα προτιμούσα να έχουμε το τσάι και να παροτρύνουμε τους διερμηνείς μας να πιούν και αυτοί ένα τσάι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας είναι η τελευταία, η λουκούμια συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και έχουμε περατώσει το νομοθετικό μας έργο γιατί φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε νομοθετικές προτάσεις. Ερχόσαστε λοιπόν σε μια τσαγκαροδευτερήτικη μέρα, σε μια παράξενη ημέρα. Παρ' όλα αυτά είμαι έτοιμος να συνεχίσω τη συζήτησή μας αύριο. Ε, έξω, συγγνώμη.